Καλημέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι άρχεται η συνεδρίαση και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη το πρώτο σημείο είναι η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Χαιρετίζω θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό τον ε, Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Δημήτρη Χριστόφια. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε και σας δίνω απευθείας το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη